Good afternoon. Καλό σας απόγευμα. Να ξεκινήσουμε παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να συγχαρώ όλους για την εκλογή ή την επανεκλογή σας και να σας συγχαρώ που επιλέξατε την θαυμάσια αυτή επιτροπή. Θα συνεργαστούμε πολύ καλά τα επόμενα πέντε χρόνια. Συγχαρητήρια για την επιλογή σας λοιπόν. Έχουμε κάλυψη από web streaming να έχετε έτοιμες τις κάρτες σας, παρακαλώ, για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Πρόκειται να συγκροτήσουμε λοιπόν το Προεδρείο με εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων. Πρώτα θα εκλέξουμε τον Πρόεδρο και μετά τους Αντιπροέδρους, λέει η προσωρινή Πρόεδρος. Η Πρόεδρος. Έχουμε λοιπόν Αντρέι Νόβακοφ από το ΕΛΚ, Σάρβαμα υπέβαλε, Νίκολας Πέξα από τους Πράσινους που αντικαθιστά Κράουβελ που αντικαθιστά Φρόιντ και Αρβανίτης αντικατάσταση του κυρίου Ομαρζή. Τώρα, οι πολιτικές ομάδες. Έχουμε από Ρινιού Καταρίντσε αντικαθιστά την κυρία Ρίτσι. Αυτά. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο προτού προχωρήσουμε τις ψηφοφορίες. Ωραία. Έχουμε απαρτία. Και θα ήθελα τις υποψηφιότητες σας για την εκλογή του Πρόεδρου. Κύριε Ντεχούφσκι αγαπητή Πρόεδρε, για Πρόεδρο της Επιτροπής, την Μόνικα Χόλμαια θα ήθελα να προτείνω, που έχει εμπειρία και συνεργάζεται ενθουσιωδώς Είναι τιμή για εμάς που την προτείνουμε για Πρόεδρο της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω Εάν η Μόνικα συμφωνεί, συμφωνώ, πρόεδρε, εκτός μικροφώνου η πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη. Επαλήθευσα ότι είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής. Έχετε συμπληρώσει και την ε, δήλωση για το οικονομικά συμφέροντα και τα δεοντολογικά. Ευχαριστώ. Αν δεν έχουμε άλλες προτάσεις θα πρότεινα να εκλέξω διαβοής. Congratulations, Monica. Συγχαρητήρια, Μόνικα, παρακαλώ να προσέλθετε, να λάβετε την έδρα. Καλή επιτυχία σε όλους για τα επόμενα πέντε χρόνια. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας και υπόσχομαι σε όλους ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ ως Πρόεδρος αν έχετε οποιοδήποτε σχόλιο, πρόταση, διαμαρτυρία αν νομίζετε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα να μου το λέτε είμαι πάντα ανοιχτή να συζητούμε τα πάντα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή για μένα. Να συνεχίσουμε τώρα με την εκλογή των αντιπρόεδρων. Μπορώ να συνεχίσω στα αγγλικά ή στα γερμανικά, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, οπω <clears throat> ήδη σημειώθηκε, έχουμε απαρτία. Δεν ξέρω αν έχουμε αλλαγές στους αναπληρωτές. Όχι. Όπως είπε και η Ματίνα, λοιπόν, Σημειώσαμε, λέει η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω τις υποψηφιότητες σας για τον δεύτερο, τον πρώτο αντιπρόεδρο. Πρόεδρε, να σας συγχαρώ και εγώ για την εκλογή σας. Κλάουντιο Μάντα, συντονιστής ε, για το S&D, προτείνω για πρώτο αντιπρόεδρο την κυρία Γαρθία Μουνιώτ. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι, Γαρθία Μουνιώτ δέχεστε την υποψηφιότητα. Será un placer, lo acepto. Βεβαίως, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είστε τακτικό μέλος της Επιτροπής μας και τα ερωτήματα που τέθηκαν και σε μένα ισχύουν και για σας. Ε, κάνατε τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και τη δήλωση που σχετίζεται με τον κώδικα κατάλληλης συμπεριφοράς. Ναι, λέτε, μάλιστα, ωραία. Οπότε θα μπορούσαμε διαβοή να κάνουμε την εκλογή. Έχει κάνει αντίρρηση, Αλλιώ μπορούμε διαβοή να εκλέξουμε την πρώτη αντιπρόεδρο. Σα συγχαίρω αγαπητοί συνάδελφοι, και σα παρακαλώ να έρθετε εδώ στο Προεδρείο. Οπότε, περνάμε στην εκλογή του δευτέρου αντιπρόεδρου. Οπότε, παρακαλώ, έχουμε ψηφιότητε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνει το λόγο. Ω σοσιαλιστική ομάδα, με μεγάλη χαρά και τιμή, προτείνω τη συνάδελφο Κατερίνα Κινίτσι. Κατερίνα Κινίτσι, λέει η πρόεδρο. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλε προτάσει. Παρακαλώ. Ο κύριο Σάλκ. Ναι. Από πλευρά ομάδα ε, I και D προτείνουμε τον κύριο Αντινόλφη. Λοιπόν, δεύτερη πρόταση. Είναι για τον κύριο Αντινόλφη. Το συνάλφα Αντινόλφη. Επειδή έχουμε δύο υποψηφιότητε, Καταρχάς, να ρωτήσω τους υποψηφίους αν δέχονται την υποψηφιότητα. Πρώτα απ' όλα κυρία Κινίτσι. Μάλιστα δέχομαι. Και κατόπιν τον κύριο Αντινόλφη. Την αποδέχομαι. Ωραία. Έχουμε δύο υποψηφιότητε. Οπότε πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματα αν έχουν κάνει τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων και τη δήλωση που σχετίζεται με τον κώδικα σωστή συμπεριφοράς. Έχετε συμπληρώσει αυτές τις δύο δηλώσεις, κυρία Κινίτσι. Ναι. Βεβαίως, στήρισα διαδικασία για όλες αυτές. Ναι, και εγώ. Έχω υποβάλει. Και εγώ τις έχω υποβάλει. Οπότε, κύριε υποψήφοι, πληρώνω τις προϋποθέσεις. Οπότε, ε, εφόσον έχουμε δύο υποψηφιότητες, θα κάνουμε μυστική ψηφοφορία όπως, ε, προτείνει, όπως προβλέπει ο ιστορικός κανονισμός. Συμφωνείτε όλοι. Να υπάρξει μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελπίζω να έχουμε τις κάρτες μας συνάδελφος και εγώ. Σε όλο τον πάρω. Λοιπόν, α κάνουμε πρώτα απ' όλα μία δοκιμή, μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Γιατί ίσω πολλοί δεν έχουν κάνει ε, ακόμη τέτοιε ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε. Γιατί έχουμε και νέα μέλη εδώ στην Επιτροπή μα. Λοιπόν, έχετε μόνο μία δυνατότητα να ψηφίσετε. Η, το ΕΛΚΑ είχε 7, οι σοσιαλιστέ 6, Renew 4, πράσινη 3, IND 3 ψήφους, ECA 3, GUE NGL 2, μη εγγεγραμμένη επίσης 2. Η εκλογή θα γίνει ως εξής. Στην πρώτη ψηφοφορία θα πρέπει ο υποψήφιος να πάρει την, την ε, απόλυτη πλειοψηφία από όσους ψηφίσουν. Στο δεύτερο γύρο εκλέγεται όποιος λάβει τις περισσότερες ψήφου. Από, όσους, ψηφίσουν τους υποψηφίου. Και αν υπάρξει ισοψηφία, εκλέγεται ο γυρεότερος. Οπότε θα πρότεινα πρώτα απ' όλα να κάνουμε μία δοκιμαστική. Δεν ξέρω αν έχετε βάλει την Μονσεράτ Καβαγέ ή τον Φιλ Κόλινς για να ψηφίσουμε. Δεν ξέρω ποιον θα ψηφίσετε. Αλλά είναι μόνο τεστ. Λοιπόν, υπενθυμίζω, αριστερά είναι το πράσινο κουμπί που εγκρίνει, το μεσαίο είναι αποχή και δεξιά είναι απόρριψη. Λοιπόν, εντάξει, εδώ η επιλογή είναι ποιος προτιμάει κρασί Δωρεάν ή ε, μπύρα δωρεάν. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγώ προτιμώ δωρεάν μπύρα. Οπότε, πέρασε. 21 ψήφοι υπέρ της μπύρας. Άριστα. Ας κάνουμε τώρα την ε, πραγματική ψηφοφορία. Με πράσινο, για αλφαβητικούς λόγους, ψηφίζεται Αντινόλφη, με κόκκινο ψηφίζεται την συνάδελφο Κινίτσι. Το καταλάβατε όλοι. Πράσινο σημαίνει Αντινόλφη. Κόκκινο σημαίνει Κινίτσι. Εντάξει, σαφές. Το καταλάβατε όλοι. Οι αποχές δεν θα λεφθούν υπόψη. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Όσο η διαρκή ψηφοφορία μπορείτε να αλλάξετε, να διορθώσετε δηλαδή την ψήφο σα από κόκκινο σε πράσινο. Όταν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία δεν μπορείτε να αλλάξετε πλέον. Λοιπόν, για όσους κάνουν λαθο Δεν γίνεται όταν κλείσει ψηφοφορία. Παραλαμβάνω. Πράσινο σημαίνει αντινόλφη, κόκκινο σημαίνει Κατερίνα Κινίτσι. Άρχεται λοιπόν τώρα η ψηφοφορία. Πέρασε. Για τη συνάδελφο Κατερίνα Κινίτσι ψήφισαν 18 συνάδελφοι. Για τον συνάδελφο Αντινόλφη 7 συνάδελφοι. Η συνάδελφος Κατερίνα Κινίτσι εκλέγεται. Sie hat die έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία. Ich darf dich, Katharina, damit bitten. Παρακαλώ λοιπόν, Κατερίνα, έλα εδώ. Οπότε περνάμε στην εκλογή τρίτου αντιπροέδρου και ζητάω προτάσεις. Από το προτείνω την κυρία Μαρτίνα Ζαμπάζοβα. Να θα κάνω σίγουρα λάθος στο Ζαμπάζοβα. Λοιπόν, Ματίνα, προτείνεσαι. Ε, υπάρχουν άλλες προτάσεις. Τότε να ρωτήσω την Ματίνα, όπως ρώτησα και τις άλλες υποψηφίου, αν έχει υπογράψει την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και τον κώδικα συμπεριφορά. Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση είναι εάν α, ε, δέχεσαι την υποψηφιότητα. Ναι. Ωραία. Μπορούμε να εκλέψουμε την συνάδελφο διαβοής. Χειροκροτήστε. Ich darf dich, Martina, bitten. Οπότε, Λοιπόν, οπότε έχουμε τέσσερις γυναίκες εδώ. Ε, πρέπει να εκλεγεί και ένας άντρας. Οπότε περνάμε στην εκλογή, αυτή για το πρόβλημα ο του τετάρτου αντιπροέδρου. Ζητώ προτάσεις. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια στις κυρίες. Πολύ θετικό το ότι θα έχουμε ισχυρές ε, γυναίκες στην Προεδρία της Επιτροπής μας και θα ήθελα να προτείνω και έναν δυνατό άντρα, Ο κύριο Ντόιτς. Ήταν εδώ στην Επιτροπή επί πέντε χρόνια, εργαστηκε σκληρά, είναι ουδέτερος προσπαθεί να βρει πάντα λύσεις και δουλεύει σκληρά πάνω στα ζητήματα αυτά. Πολέμησε τη διαφθορά σε πολλές χώρες και θα ήθελα να τον ψηφίσετε. Άλλες προτάσεις υπάρχουν. Όχι. Να ρωτήσω τον κύριο Ταμαστούιτση αν Ναι, ναι, έρχομαι σε εσά. Δέχεστε την υποψηφιότητα. Ναι. Και έχει υπογράψει την δήλωση οικονομικών σφαιρόντων και τον κώδικα συμπεριφορά. Ναι, ναι, έχω υποβάλει όλα τα έγγραφα. Να δώσω τον λόγο στον συνάδελφο κύριο Μάντα. Ε, ε εξ ονόματος των σοσιαλδημοκρατών θα θέλαμε μυστική ψηφοφορία για αυτήν την υποψηφιότητα. Ζητήθηκε μυστική ψηφοφορία. Θα έχουμε λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία. Χρειάζεται πάλι τεστ. Πρώτα απ' όλα, ποιος συμφωνεί με το αίτημα για μυστική ψηφοφορία. Πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι βουλευτές. Αλλιώ δεν θα είναι μυστική η ψηφοφορία. Είναι πάνω από έξι βουλευτές από ό,τι βλέπω. Οπότε θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ωραία. Ποιο? Μάλιστα, το πράσινο κουμπί σημαίνει ότι ψηφίζεται υπέρ του υποψηφίου, το κόκκινο κουμπί κατά. Οι εποχές δεν θα μετρήσουν. Θέλετε να κάνουμε ένα τεστ πάλι, όχι. Ωραία. Ε, να προσθέσω πως ε, τα λάθη μπορούν να διορθούν μόνο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και όχι μετά. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έντεκα υπέρ, 6 κατά. Τρεις αποχές, δεν μετράνε. Ε, επί 20 ψήφισαν Οπότε, ο συνάδελφος συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία. Τάμας, παρακαλώ. Ας έρθει και ένας άντρας στο Προεδρείο.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 Και βεβαίως ε, σίγουρα θα εργαστούμε εντατικά γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα που θα μας απασχολήσουν και οπωσδήποτε με τις και τους ε, συμπροέδρους εδώ πέρα θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στην ε, κληρονομιά, στην πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στο παρελθόν σε αυτήν την Επιτροπή. Πάντα θα έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, θα είμαστε στην διάθεσή σας. Ε, το κινητό μου είναι στην διάθεσή σας εάν υπάρχουν προβλήματα. Και νομίζω ότι Βεβαίω, συγχαίρω και τις ε, αντιπροέδρους ε, και τον αντιπρόεδρο. καλό απόγευμα σας εύχομαι. 24 Ιουλίου είναι η πρώτη μας συνεδρίαση και θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την επιστημονική μας υπηρεσία στην διάθεσή μας. Θα περάσουμε κατευθείαν στην δουλειά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ε, πειθαρχία. Τα λέμε τότε.